ο εκπροσωπός πρόεδρος του. Και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο. Για το πώς δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει να συνεργαστεί με την ε, ε, Προεδρία 2,5 ετών όσον αφορά την χρονική διάρκεια από πλευράς ε, Προεδρίας και πώς προβλέπει να συνεργαστεί με την ανακυκλούμενη Προεδρία. Η εκπεριτροπής ανακυκλούμενη Προεδρία, σε αυτή την περίπτωση τώρα η Ισπανική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της για τους επόμενους έξι μήνες, πάντα φυσικά στις αρχές αυτής της περίοδου έξι μηνών όπως σήμερα και θα υποβάλει και μία μια τελική έκθεση κατά τα τέλη του εξαμήνου. Η Προεδρία, η διαρκή η σταθερή Προεδρία του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του, της ε, Συνόδου. Κάθε ε, ε, έτος έχουμε δύο Συνόδους και έτσι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των Συνόδων Κορυφής δύο φορές δηλαδή αναεξάμεινο, τέσσερις φορές αναέτος δηλαδή. Αυτά είναι όλα όσα είχα να αναφέρω σε σχέση με ε, πληροφορίες που ήθελα να σας δώσω και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου παρουσίαση του προγράμματος της Ισπανικής Προεδρίας. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ισπανικής Κυβέρνησης, ε, τον κύριο Θαπατέρο που είναι ο προεδρεύων της εξάμηνης ε, Προεδρίας.